annoncé. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Άρχεται η σημερινή συνεδρίαση. Να ξεκινήσουμε μία μικρή ανακοίνωση. Χθες αποφάσισε η συνέλευση